I would ask the colleagues to take their seats because we... would... Παρακαλώ καθίστε αγαπητοί συνάδελφοι να ξεκινήσουμε συντόμως με τις ψηφοφορίες. So, when Mr. Liberatsky will get to his place... Όταν καθίσει και ο κύριος Λιμπεράτσκι θα ξεκινήσουμε. În regulă. Deci, prima chestiune pe care trebuie să o lămurim ένα θέμα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αρχικά. Πρακτικά, παρακαλώ, Κάρβα, έχετε να έτοιμα επί της διαδικασίας. Thank you, Mr.